Πολλές φορές ε, οι συζητήσεις είναι πολύ βαρετές, ε, αλλά τώρα ήταν πολύ πιο ζωντανή. Σας εύχομαι λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε.